αποτελεσματικά αποφάσεις προς το συμφέρον των πολιτών της Ένωσης. Αυτές ήταν οι ανακοινώσει του Προέδρου. Τα δε πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα έχετε στη διάθεσή σα. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Οπότε θεωρείτε πως τα πρακτικά εγκρίνονται. Κυρίες και κύριοι. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Μάρο. Yeah. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρωί στο Αφγανιστάν δύο Ιταλοί στρατιώτε, της στρατιάς του Ρινέντς ε, σκοτώθηκαν από μια απόπειρα παίζει, προσπαθεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την καταπολέμηση του πολέμου. Θα ήθελα κατά τη συνόδου να απευθύνει σε λυπητήρια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων που περνούν πολύ δύσκολες στιγμές. Ε, ε, ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ο κύριος Πιτέλα έχει ζητήσει τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ζητάω ενός λεπτού αγόρευση, χρόνο αγόρευσης για να εκφράσω και εγώ τα ίδια πράγματα που εξέφρασε ο συνάδελφος κ. Μαόρο με τον οποίο ε, συμφωνώ και απευθύνω και εγώ προς τα συλληπιτήρια που θέλει να απευθύνει ο κ. Μαόρο και νομίζω ότι όλη η Ολομέλεια θέλει να απευθύνει τα συλληπιτήρια για αυτούς τους δύο Ιταλούς στατώτους που σκοτώθηκαν στην πρωινή απόπειρα σήμερα. Θα πρέπει και καταδίκη και αλληλεγγύη μαζί με τα συλληπιτήρια πρέπει να πάει προς την οικογένεια ε, θα πρέπει να καταδικαστεί κάθε μορφή τρομοκρατίας αλλά και μια ανανεωμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δίπλα στα κράτη-μέλη, στη δράση του κατών μελένων, ούτως ώστε να πιο αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές και να υλοποιούνται και να λαμβάνουν χώρα σε μια κατάσταση μεγαλύτερης ασφάλειας ειρηνευτικές αυτές προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Κύριε Πιτέλα. Και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο κυρίους που μας επέστησαν την προσοχή πάνω σε αυτό το γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε αυτές τις πράξεις βίας που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες οι οποίοι είναι σε ενεργό υπηρεσία στο Αφγανιστάν εκ μέρου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ήθιστε εμείς να αναλύουμε και να σκεφτόμαστε αυτές τις στιγμές αυτά τα γεγονότα. Κύριος Βανόρντεν, κύριε Πρόεδρε, ενώ σκεφτόμαστε και θυμόμαστε τραγικές απώλειες στο Αφγανιστάν, θα έπρεπε επίσης να θυμηθούμε ότι σχεδόν καθημερινά χάνουμε Βρετανούς στατιώτες που δίνουν τη ζωή τους σε αποστολή του ΝΑΤΟ που και αυτή πραγματοποιείται σε αυτή τη χώρα. Βεβαίω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την τραγική απώλεια, τι τραγικέ απώλειε και απευθύνουμε την ιδιαίτερη συμπάθειά μα προ τι οικογένειε όλων των στρατιωτών, ανεξάρτητα από ποια χώρα ε, υπηρετούν υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ εκεί. Συμφωνώ, λέει ο Πρόεδρο, συμφωνώ απολύτω μαζί σα με την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Βανόρντεν Όλοι νομίζω ότι έχουμε παρόμοιες απόψεις. Είναι Ευρωπαίοι οι οποίοι βοηθούν όλους μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της βίας στον κόσμο, εκπροσωπούν όλους μας. Ο κύριος Χένεν. Είναι φυσιολογικό να αποτείουμε φόρο τιμή σε όσου χάνουν τη ζωή του ε, επί το έργο. Θα ήταν επίση ε, χρήσιμο να σκεφτόμαστε και τους ε, ε, μισθωτούς ε, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους ε, πολύ συχνά κάθε μέρα επειδή οι εργοδότες τους δεν θέτουν στη διάθεσή τους τα μέσα που χρειάζεται για να προστατεύσουν τη ζωή τους στον χώρο εργασίας. Κυρίες και κύριοι, έχω να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα σημαντικό θέμα.